darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε. την ε, επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί στις 23 Ιουνίου 2016. Σε απόλυτη συμφωνία με τις ε, πολιτικές ομάδες